Ευχαριστώ Επίτροπε. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον προγραμματισμό των διαστατικών ταμείων για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και υποστήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συγχωρείτε, για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω λέγοντας ξανά πως δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη και η τελευταία σύνοδος παραδέχτηκε αυτό το οποίο λέγαμε εμείς εδώ πέρα πισματικά εδώ και χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη λιτότητα πρέπει να είναι φιλική για την ανάπτυξη. Οι προβλέψεις δεν είναι καλές. Από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούμε σε διάβρωση του παραγωγικού δυναμικού, ειδικά του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης και ειδικά των νέων. Οπότε θα πρέπει να καταβάλουμε όλοι οι προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης για να εκμεταλλευτούμε τον ευρωπαϊκό προεπιλογισμό. Στο πλαίσιο αυτό μας εξέπληξε το ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως υπάρχουν 82 δισεκατομμύρια ευρώ αδιάθετα όπως τα είπε στα διαρθρωτικά ταμείο, 22 δισεκατομμύρια στο κοινωνικό ταμείο, που είναι γύρω στο 30% του ποσού του 2007-2013 και 60 ε, εκατομμύρια στο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μεγάλο ποσοστό δηλαδή του προϋπολογισμού. Αλλά ανακαλύψαμε πως δεν είναι κονδύλια τα οποία δεν έχουν ξοδευτεί, αλλά δεν έχουν ξοδευτεί ακόμα. Κοιτώντας δε προσεκτικά την ανακοίνωση, αντιλαμβανόμαστε πως δεν έχουν διατεθεί ακόμα σε συγκεκριμένα έργα, αλλά έχουν δεσμευτεί ναι. σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πως η κατανομή σε έργα μέσω διαγωνισμών είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί μέχρι το τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών. Άρα μπορούμε να αναμένουμε πως τα περισσότερα κράτη-μέλη θα κρατήσουν ένα κομμάτι Τη κατανομή αυτή για το 2012 και 2013. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πως το υπόλοιπο 70% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχή είτε ήδη έχουν εκταμιευθεί είτε έχουν υποβληθεί προσφορές, άρα υπάρχουν ήδη νομικές δεσμεύσει. Το ερώτημα μας λοιπόν είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως από την Κομισιόν την η δυνατότητα αναπρογραμματισμού. Αντιλαμβανόμαστε πως ε, βεβαίως ε, είναι προτεραιότητες ούτως ή άλλως οι θέσεις εργασίας από το 2007 και μετά όσον αφορά την πολιτική συνοχή, αλλά συμφωνούμε πλήρως πως η δυνατότητα της πολιτικής συνοχής για να δημιουργεί θέσεις εργασίας πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Αυτό το οποίο όμως είναι ενισχυτικό είναι πως ο πιθανός αναπρογραμματισμός αυτός της κατανομής των κονδυλίων στα τελευταία δύο χρόνια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη, μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες ερμηνείες και έτσι να υποβαθμίσει την εικόνα της πολιτικής και της πραγματικού της αντικτύπου. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε όλες τις προτάσεις της Κομισιόν που στόχο είχαν να ενισχύσουν την αντίδραση στην κρίση. Σε χρόνο ρεκόρ υιοθετήσαμε τροπολογίες στο Γενικό Κανονισμό για να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό με τον οποίο θα μοιραζόμαστε τον κίνδυνο για τη διευκόλυνση χρήση των κονδυλίων σε χώρε που το έχουν ανάγκη. Οπότε να πω πως βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν προβλήματα απορροφητικότητα σε κάποιες χώρες και Εκτιμούμε τις ε, προσπάθειες κομισιών να βοηθήσει χώρες όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Ελλάδα να βγουν από την παγίδα αυτή της λιτότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των διατροφικών ταμείων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, η οποία μα δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το πιο δυναμικό υπάρχει για ανάπτυξη στην περιφερειακή πολιτική παρά το ότι γνωρίζω πως εξορισμού βεβαίως πράγματι πάντα προσανατολισμένη ήταν στην ανάπτυξη η πολιτική συνοχής. Παρόλα αυτά πολύ περισσότερο τώρα σε καιρούς τέτοιους θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην ανάπτυξη. Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την ύφεση την οποία αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Το πρώτον είναι η προώθηση και η ενίσχυση των μικρομεσαίων εγχειρήσεων και δεύτερον η εξαιρετικά υψηλή ανεργία των νέων που σε κάποιες χώρες φτάνει το 50%. Χρειαζόμαστε λοιπόν να πρέπει να στηρίξουμε και τους δύο τομείς αυτούς. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε 23 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και 23 εκατομμύρια επίσης ανέργους. Εάν απλά να σας το πω κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάβει έναν άνεργο, το πρόβλημα της ανεργίας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου αποφάσισε πώς θα εστιαστεί ακόμη περισσότερο η διαρθρωτική πολιτική στην ανταγωνιστικότητα για να υπάρξει έτσι ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα χωρίς ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρότειναν οτιδήποτε δεν έχει πάει σε συγκεκριμένο έργο πράγματι ε, σωστά μιλήσατε για 22 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ε, ανάλογα ποσά από το ΕΤΠΑ να πάνε στην βέλτιστη χρήση ή τουλάχιστον να επανεξεταστούν για να δούμε ποια θα είναι αυτή η βελτιστή κρίση. Και πράγματι, επί της αρχής έχουν ήδη διατεθεί σε προγράμματα, αλλά όχι σε συγκεκριμένα έργα τα ποσά αυτά. Γι' αυτό νομίζω πως μπορούμε πράγματι θεμητά να πούμε, να δούμε ακόμη μία φορά, μήπως μπορεί να υπάρξει μία βελτίωση των δομών και οι Κομισιόν προσφέρθηκε να βοηθήσει κάποιες χώρες με την εμπειρία την οποία έχουμε, ειδικά όσον αφορά το πρόβλημα της ε, υψηλής ε, ανεργίας ε, των νέων, γιατί σε τόσο κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να μας επιτραπεί να εξατλήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και είμαστε στην διάθεση των κρατών μελών. Κάναμε αυτή την προσφορά, τα κράτη-μέλη την δέχτηκαν τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, συνομιλίες ε, αρχές Μαρτίου, αλλά όπως σας είπα επαφίεται στα κράτη-μέλη το εάν θα προσαρμόσουν τα προγράμματά τους. Όπως είπα, για τους στόχους αυτούς, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με βάση αυτά λοιπόν, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που έχει επιδείξει για να έχουμε γρηγορότερα τη λήψη μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας να τα ξεπεράσουμε και να ολοκληρώσουμε έργα. Και τέλος, όπως είπα, είμαστε έτοιμοι όπως κάνουμε μέρα τη μέρα να κάνουμε μία προσαρμογή, μία ρύθμιση εάν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν είναι έτοιμη, αλλά ζητάω και τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας βοηθήσετε κι εσείς για να καταπολεμήσουμε, όπως είπα, την ενεργεία των νέων και να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε τώρα οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κ. Βαν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απόψινή παρέμβαση βεβαίως έχει στόχο να καταστήσει τα πράγματα ε, σαφή και πράγματι η κυρία Χίμπνερ ήθελε να μάθει τι, ε, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να απελευθερώσει 22 δισεκατομμύρια ευρώ για τους στόχους που αναφέρατε. Αυτά δεν ε, πριν από μια μισή εβδομάδα είχατε έρθει επίσκεψη σε εμάς στην Ολλανδία. Και τι μας είπατε, υπάρχουν εταίροι, ε, δίνεται τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ε, αναζητείτε πανεπιστήμια, εταιρείες, περιφέρειες για να δεσμεύσουν άλλα 3-4 ευρώ. Και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Δηλαδή ο προγραμματισμός απαιτεί χρόνια δεν μπορεί να ανατραπεί. Ποια είναι η εμπιστοσύνη που μπορούν να δείξουν μετά όλοι αυτοί οι φορείς. Γιατί, να σας πω, τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε, είναι ένα λογιστικό κόλπο άρα ή μπορεί ανά χώρα να δοθεί, το έχετε δοθεί και υπάρχει συγκεκριμένο ποσό για Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι πως σε, την επόμενη μέρα στις ε, εφημερίδες γράφανε ε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με έργα τα οποία δεν θα γίνουν ε, με τα διαρθρωτικά ταμεία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ποια είναι τα περιθώρια, ποιο, εντός ποιανού πλαισίου κινείστε ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Κρέλ για 3,5 λεπτά. Κυρία Κρέλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τρία πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν ε, ασχολείται επιτέλους με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Δεύτερον, χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν βλέπει πως ακριβώς σε καιρό κρίσης δεν μπορούμε να έχουμε μόνο σκληρή λιτότητα αλλά και επενδύσεις χρειάζονται και βεβαίως ε, στην πρώτη γραμμή είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί αυτές δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Τρίτον, ρωτάω ξεκάθαρα, όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ, ο κύριος Μπαρόζο δημιούργησε την εντύπωση πως μπορεί να εμφανίσει 82 δισεκατομμύρια ευρώ λεφτά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και δημιουργείται εδώ πέρα η αίσθηση πως δεν χρησιμοποιούνταν σωστά αυτά τα παράγματα στην πολιτική συνοχής. 82 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα μιλάμε σχεδόν για ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής μέχρι το 2013. Από όσο ξέρω όμως έχει ενταχθεί σε προγράμματα και δεσμευτεί σε συγκεκριμένα έργα το ποσό αυτόν. Πώς θα το οργανώσετε να πούν όλες οι περιφέρειες ναι εντάξει θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό και επειδή εμείς δεν έχουμε τόσο ψηλή ενεργεία των νέων να πάνε τα λεφτά σε άλλες χώρες. Αναμένω ειλικρινά σας λέω την αντίδραση γιατί ενοχλήθηκαν οι περιφέρειες. Έρχονται σε μένα και μου λένε μα τι γίνεται τώρα να μας πάρουν τα λεφτά. Και εδώ πέρα θέλω να σας αποτρέψω η πολιτική συνοχής είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Είναι αυτή η οποία είναι πιο ορατή και πιο απτή για τον πολίτη και δημιουργεί εμπιστοσύνη. Και αν τώρα κάνουμε τέτοιες ε, δηλώσεις γενικές ε, ότι θα δώσουμε τα λεφτά από εδώ και από εκεί, δημιουργείται η εντύπωση πως ε, μπορούμε να βρούμε από εδώ και από εκεί κάτι δισεκατομμύρια. εκατομμύρια αυτά τα πράγματα δημιουργούν αβεβαιότητα και αν σκεφτούμε πως το Συμβούλιο για τις ε, φετινές διαπραγματεύσεις δεν θα εγκρίνει τις δαπάνες που ζητάει η Κομισιόν και Κοινοβούλιο και μιλάμε για έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ε, και κοστίζουν 15 δισεκατομμύρια και τελικά θα βρεθούν με 5 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Αν ρωτιέμαι πώς μπορούμε να δημιουργούμε την εντύπωση πως τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να πληρώσουν περισσότερα λεφτά για την πολιτική συνοχή. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ε, πράγματι να ασκήσουμε τη σωστή πολιτική, να υποστηρίξουμε τις χώρες με την ψηλή ανεργία των νέων, αλλά δεν πρέπει να δημιουργούν περισσότερη ανασφάλεια σε δύσκολους καιρούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την Άλντε. Μανέσκου για δύο λεπτά. Ε. Κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναπρογραμματισμό των πόρων που δεν έχουν κατανεμηθεί προς την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καταπολέμηση ενεργείας των νέων είναι κάτι ευπρόσδεκτο, κυρίως εφόσον έχει τονώσει, τονίσει ιδιαίτερα το πρόβλημα οικονομική κρίση. Για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υψηλό επίπεδο απορροφήσεω ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να αποφασίσουν ποιε είναι οι προτεραιότητες του όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Ξέρετε ότι δεν είναι το πρώτο μέτρο κατά της κρίσεως αυτού του είδους. Η κυβέρνηση της χώρας μου, που ίσως έχει τις ε, μικρότερες επιδόσεις όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων, η εμπειρία της χώρας μου δείχνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντα σωστά αυτοί οι πόροι. Η απορρόφηση εξαρτάται και από τις εθνικές κυβερνήσεις που πρέπει να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις τα μέτρα αυτά και να πετύχουν καλά αποτελέσματα. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σας έθεσε η Επιτροπή ε, Ρέτζη και να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Να μας πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες έδειξαν ότι δεν εφαρμόζουν τα μέτρα αντικρίσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλά και πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι κυβερνήσεις θα χειριστούν σωστά τα χρήματα που τους διατίθενται ώστε να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί η ενεργεία των νέων. Ε, ε, αναφέρθηκε και αναφέρεται κάποιες χώρες όπου η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ ψηλή. Στη Ρουμανία ε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ πραγματικό. Οι Ρουμάνοι οι υπήκοοι θέλουν να ξέρουν κατά πόσο θα πάνε για άλλους σκοπούς τα χρήματα τα οποία είχαν διατεθεί αρχικά για τη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Σρέτερ για 1,5 λεπτό. Κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω το ότι το Συμβούλιο ακολούθησε τη Συμβουλή του Κοινοβουλίου και θέλει να καταπολεμήσει την Ανοιγία των νέων. Και αυτά τα οποία πρότεινε ο κύριος Μπαρόσο, η λεγόμενη εγγύηση για τους νέους, ήταν πράσινη πρόταση. Σε πράσινη έκθεση πρωτοβουλία. Σε αντίθεση όμως με τον κύριο Μπαρόσο, εγώ θέλω να δοθεί ιδιαίτερο βάρος μειονεκτικού νέους. Και γι' αυτό χρειάζεται αποκεντρωμένη δράση. Αυτή είναι η καλύτερη. Τα λεφτά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να παραμείνουν επί τόπου και εκεί πέρα να χρησιμοποιηθούν. Αυτά προς τον κύριο Μπαρόσο. Η ομάδα μας υποστηρίζει επίσης την απόφαση του Συμβουλίου για την πράσινη οικονομία. Επίσης πράσινη έκθεση ήταν που πριν από δύο χρόνια εγκρίθηκε στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία. Γι' αυτό αυτό το οποίο ζητάμε για ένα προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων εκεί όπου χρειάζονται πρωτοβουλίες για την πράσινη οικονομία. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μία τέτοια γραμμή έχει ουσιαστική σημασία γιατί τότε θα είναι ανταγωνιστικές. Δεν μιλάμε απλά για να αλλάζουν τα παράθυρα, αλλά έργα από τα οποία θα μπορούν να αποφεληθούν οι επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ ο Μαρζή για δύο λεπτά εκ του. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι λογικό να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη για νέα ανάπτυξη πόρων, ενώ το Κοινοβούλιο να βρίσκεται αποτελεσμένου. Μας λένε ότι 82 δις ευρώ δεν καταναλώθηκαν και ούτε και θα καταναλωθούν μέχρι το 2013. Τελικά τι μας ζητούν, να σας πιστέψουμε, να πιστέψουμε αυτά που λέτε. Εγώ όμως θέλω να καταλάβω, να τα δω τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Πώς μπορείτε βέβαιοι να είστε ότι το 2012 δεν θα πανηθούν οι πόροι αυτοί, πριν δηλαδή το τέλος της περίοδου προγραμματισμού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμία περιφέρεια που αρχικά ήταν δικαιούχος των κονδυλίων αυτών δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί ουσιαστικά με την αυτή ανάπτυξη πόρων. Και τελικά, Ποιος είναι ο λόγος αυτής της ε, νέας ανάπτυξης πόρων, μήπως είναι κάποιος άλλος ο λόγος, μήπως δηλαδή τελικά θέλετε να μετριάσετε τα καταστροφικά αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας, τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μετριάσετε τα αποτελέσματα της κρίσης, δεν θα ήταν πολύ πιο σκόπιμο και καλό να κινητοποιήσετε νέους πόρους να κινητοποιήσετε λοιπόν νέους πόρους για να χρηματοδοτήσετε πραγματικές πολιτικές ανάπτυξης και πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων. Και ενώ το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που εδώ και πολύ καιρό ζητούμε αλλά που εξακολουθεί να μην έχει αποκρισταλωθεί σε συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους άλλους εγγεγραμμένους αγορητές. Θα δώσω το λόγο. Ε, Τσέλερ για δύο λεπτά. Κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Προξενεί εντύπωση το ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς τι είναι διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής. Είναι εξορισμού η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναγκαιότητά της έχει ήδη αποδειχτεί στον καιρό της κρίσης. Βεβαίω, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την ανάπτυξη των επιχειρησιακών αυτών προγραμμάτων γίνεται όπως περιγράφεται στα σχετικά προγράμματα. Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη και περιφέρειες συνεργάζονται και έτσι δημιουργούν μια πραγματική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Η επιτυχία λοιπόν αυτής της πολιτικής βασίζεται στην αξιοπιστία των προγραμμάτων αυτών και των κονδυλίων που έχουν προϋπολογιστεί. Γι' αυτό απορώ πως Κομισιόν και κράτη-μέλη προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική συνοχής για πάσα νόσο. Δεν είναι σωστό αυτό και επιπλέον οδηγεί τους φορείς στις διάφορες περιοχές οι οποίοι έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμο προγραμματισμό σε αβεβαιότητα. Οπωσδήποτε είναι σημαντικός ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης ανεργίας των νέων, αλλά αυτό θα γίνει αν διατηρηθούν οι εταιρικές σχέσεις και συμφωνίες μεταξύ Ένωσης Κομισιών Κρατών Μελών και Περιφερειών γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν το τι χρειάζεται στην κάθε περιφέρεια. Και έτσι θα πρέπει να υπάρξει και αυτή η αλληλεγγύη η οποία καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση ορατή στις περιφέρειες και θα πρέπει έτσι εύκολα να την ξεχνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Η Η Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι χωρίς νέους δεν υπάρχει μέλλον. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι με τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε λύσεις. Λύσεις που δεν θα έλθουν ε, εάν ε, στηρίξουμε εργασιακές μεταρρυθμίσεις ε, σαν αυτές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μου που κάνει πιο επισφαλή την εργασία. Η Ευρώπη έχει γύρω στο 23% των νέων ανέργου. Στη χώρα μου την Ισπανία 49% των νέων είναι άνεργοι. Πολύ περισσότεροι, πολύ μάλλον από αυτούς είναι ε, με υψηλή μόρφωση, οι οποίοι δείχνουν τελικά ότι πλέον έχουν μπουχτήσει, έχουν κουραστεί ε, που δεν βλέπουν να υπάρχει λύση. Πρέπει να βρούμε λύση, να βοηθήσουμε να προσλαμβάνονται νέοι, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίω αυτές που ε, δημιουργούν νέοι. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ προτεραιότητα η εκπαίδευση να είναι προσαρμοσμένη στην αγορά εργασίας δηλαδή να είναι πιο ισότιμο, πιο δίκαιο το σύστημα της εκπαίδευσης που θα καταργεί διαφορές μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και έτσι θα τονωθεί η δημιουργικότητα, η καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα, η δίκευση και η κινητικότητα των σπουδαστών. Η Κομισιόν μπορεί να μας εξηγήσει πώς θα κατανεμηθούν μεταξύ των διαφορετικών ταμείων τα ποσά τα οποία θεωρεί ότι θα δοθούν στην Ισπανία, ότι αντιστοιχούν στην Ισπανία και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από τα 82 δι ευρώ που δεν έχετε ακόμη επιμεριστεί ε, και θα πάνε σε αυτό το ταμείο. Τι θα γίνει συγκεκριμένα με την Ισπανία, ποιο θα είναι το ποσοστό που αναλογεί στην Ισπανία. Τέλο, η Κομισιόν πώ θα ε, συμπεριλάβει τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ καθώ ε, και του κοινωνικού εταίρου στα σχέδια δράση. Ελπίζω κύριε Επίτροπε να έχουμε γρήγορα ε, μια αποφασιστική βιώσιμη λύση διότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία μέρα ακόμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Τέρερ. Κύριε Στέρερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν πρωτοβουλία των φιλελευθέρων η επισήμανση αυτή πως ε, δηλαδή είναι χαμηλά τα ποσοστά απορροφητικότητας και την έκθεση είπαμε που βρίσκονται οι αιτίε. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να δραστηριοποιηθεί και την υποστηρίζουμε στις προβληματικές χώρες ε, στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, στην Νότια Ιταλία να πάνε αυτά τα κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση των νέων, στην ανεργία των νέων, οπωσδήποτε και αποφασιστικής ε, σημασίας είναι βεβαίως και η δυνατότητα των κρατών μελών να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά η εντύπωση που έχουν οι πολίτες, όπως στην Ελλάδα, είναι πως τα πράγματα δεν λειτουργούν. Η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί και η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αποφασίζει μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζει. Οπότε το πρόβλημα. Τι είναι, είναι σαν να πατάμε τον γκάζι σε ένα αυτοκίνητο και να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού σε όλο αυτό το μηχανισμό της ε, μετάδοσης χάνεται η επαφή με την πραγματική οικονομία για να καταπολεμήσουμε το ζήτημα στη ρίζα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Μιράντα για ένα λεπτό. Κυρία Μιράντα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κύριε Επίτροπε, έχει τους ε, πιο καλά εκπαιδευμένους ε, νέους που είναι πιο καλά προετοιμασμένοι από οποιονδήποτε άλλο καιρό, αλλά δυστυχώς μια νεολαία που πλήττεται από την ανεργία και οι θέσει εργασία είναι πάρα πολύ κακές. Αυτή τη στιγμή συζητούμε τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Ο δείκτης ε, ανεργίας και συγκεκριμένα των νέων μπορεί να είναι ίσως ε, και ένας από τους επόμενους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το εισόδημα. Σε χώρες όπου οι νέοι κάτω των 25, η μισή τουλάχιστον είναι άνεργοι. Τι μέλλον έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε σταθερές συμβάσεις, ε, Θέλουμε δίκαιους μισθούς, αντίθετα με αυτά που προτείνουν κάποια κράτη, όπως και η Ισπανία, που έκανε μια αντικοινωνική εργασιακή, εργατική μεταρρύθμιση. Έχουμε λοιπόν τόσο καλά εκπαιδευμένους νέους. Τι τους προσφέρουμε, κακές θέσεις εργασίας, μερική απασχόληση, ανεργία, ακόμη και ε, τη μετανάστευση ως επιλογή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημο άλοθη η κρίση για να περάσουν εργασιακές μεταρρυθμίσεις που τελικά προτείνουν ε, και επιβάλλουν λιτότητα. Και σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έκλεισαν. Έβαλαν Λουκέτο ακριβώς λόγω αυτής της κρίσης. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ernst, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, κύριε Ernst, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εκπλήσω με κάπως αφού πέρασε ο κ. Μπαρόσο και οι συνάδελφοί του του Συμβουλίου χρόνια πέρασαν εξετάζοντας αυτές τις πολιτικές για να καταπολεμήσουν την ανεργία. Και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι η κρίση δημιούργησε μεγαλύτερη ανεργία. Βλέπετε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται συζήτηση για περισσότερους πόρους. Και ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα λεφτά που θέλετε να διατεθούν. Ψηλά θα έλεγα, πλησιάζουμε το 2013 και ήδη έχει γίνει ο προγραμματισμός. Ξέρετε όμως πως αυτά τα πράγματα έχουν ήδη δεσμευτεί. Μην κάνετε κολπάκια. Τι γίνεται με την Ιρλανδία, θα επαρκέσουν ε, τα κονδύλια. Οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει τα κονδυλιά τους. Τι θα του πείτε εκεί πέρα για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Ναι, κυρίε και κύριοι, χρειαζόμαστε όθηση στην πολιτική της απασχόληση, ειδικά για τους νέους, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά υπαρκτά λεφτά. Και χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, μια λογική προστασία από τις απολύσεις και αξιοπρεπή εργασία. Και θέλω να πω επίσης το τι δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο μακροοικονομική αιρεσιμότητα και θα πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να μας πείτε τι σημαίνουν αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ. Λουκατσεύσκα, για δύο λεπτά. κυρία Λουκατσεύσκα έχει λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η οικονομική κατάσταση και η ψηλή ανεργία των νέων ζητούν ε, κατεπίγουσα δράση. Γι' αυτό χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος αυτής, ο κ. Μπαρόσο, παρατήρησαν αυτό το πρόβλημα και θέλουν να αναπρογραμματίσουν τα διευθυντικά ταμεία και να θέσουν πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν την ενεργεία των νέων. Ερώτηση, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με, αποδοτικά, με αποδοτικό τρόπο, ομαλά και γρήγορα και 82 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο είναι πράγματι διαθέσιμα. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να κάνουν ένα προγραμματισμό των διαθροτικών ταμείων διότι σήμερα πάνω από το 20% των νέων στην Ευρώπη ε, βρίσκεται στην ενεργεία ε, κατά μέσο όρο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την καταπολέμηση της ενεργείας όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν τα μη δαπανηθέντα ποσά αλλά να δαπανηθούν αποτελεσματικά. Είναι σημαντικό ε, τα ευρωπαϊκά ποσά που διατίθενται για την κατάρτιση να παρέχουν υψηλή ποιότητα κατάρτιση που θα δίνουν τι δεξιότητε που είναι αναγκαίε για την αγορά εργασία. Αυτό που είναι σημαντικό για τι νέε θέσει εργασία είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα έπρεπε να είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μόνο 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ηγούνται στην καινοτομία. Πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θέλουν να ζητήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση διότι είναι πολύ μακρά η διαδικασία ε, είναι επαχθής και δεν είναι σαφής. Όλοι συμφωνούν ότι η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον και η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του ΑΕΠ, για την καταπολέμηση ανεργία και για την επίτευξη οικονομική σταθερότητα. Νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι για τη σημερινή συζήτηση ε, ξέρουμε ότι χιλιάδε άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουν κάποια μέτρα. Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα λοιπόν. Πώς συγκεκριμένα βλέπετε ότι θα πετύχετε την υποστήριξη των μικρομεσών επιχειρήσεων. Πώς θα καταπολεμήσει την ενεργεία των νέων συγκεκριμένα και πώς θα είναι αποτελεσματική η προσπάθεια. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ουλσκογ για 1,5 λεπτό. Κυρία Ουλσκογ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της οικονομική κρίση στην Ευρώπη είναι το υψηλό επίπεδο της ανεργίας των νέων. Κάποιοι αγορητές είπαν ότι σε κάποιες χώρες φτάνει και το 50% η ανεργία των νέων. Ήδη στις εκλογές του 2009 ο πρόεδρος Μπαρόσο είχε υποσχεθεί ότι η καταπολέμηση της των νέων θα ήταν η απόλυτη ύψιστη προτεραιότητα της θητείας αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως μέχρι τώρα δεν είδαμε πολλές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσει ε, για να γίνει κάτι. Διότι εδώ δεν ασχολούμεθα με, τις, ε, με τους νέους και το μέλλον των νέων. Φαίνεται να διαφορούμε. 100 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται διαθέσιμα. Θα ήταν φανταστικό αν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Είναι αργά, είναι πάρα πολύ αργά. Λέει είναι κατεπήγον να κινηθούμε, να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, διερωτώμεθα, γιατί αυτά τα χρήματα πρέπει να αφαιρεθούν από τα ιδιωτικά ταμεία. Η πολιτική της συνοχής δεν θεωρείται προτεραιότητα. Υπάρχουν και άλλα κονδύλια του προπολογισμού στα οποία θα έπρεπε να προσφύγουμε αντί να πειράξουμε τα διεθνωτικά ταμεία. Και πόσο χρόνο, πόσο χρόνο θα χρειαστούμε ούτως ώστε να διατεθούν αποτελεσματικά αυτοί οι πόροι, να καταβληθούν τα ποσά. Είναι κατεπήγον θέμα για τους νέους. Θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα για τους νέους. Ευχαριστώ. για ε, ένα λεπτό. υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική συνοχή εδώ την ίδια στιγμή προωθείται μια πολιτική με ευθυνική της κομισιόν η οποία οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας και σε κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελλάδα. ξέρετε ότι σήμερα η ανεργία μεταξύ των νέων στην ελλάδα έχει φτάσει στο 48% και το γενικό σύνολο της ανεργίας στον πληθυσμό είναι 20,9% και μάλιστα με το νέο μνημόνιο εξαναγκάζονται οι νέοι κάτω από τα 25 να δουλεύουν με μειωμένο μισθό κατά 32% και επομένως ένας νέος 25 ετών να εισέρχεται στην αγορά εργασίας με μισθό 440 ευρώ για οκτάωρη απασχόληση σε ένα ολόκληρο μήνα. Με αυτές τις συνθήκες βέβαια οι νέοι τείνουν να φύγουν από τη χώρα υπάρχει πράγματι μια πολιτική που να έχει συνοχή δηλαδή αυτές οι πολιτικές που συζητάμε εδώ πέρα για κοινωνική συνοχή για απασχόληση των νέων συνάδουν με τα μέτρα που προωθούνται μέσα από το, νέο μνημόνιο. εδώ είναι μεγάλο το θέμα. υπάρχουν αδιάθετοι πόροι πράγματι μπορούν να στραφούν για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για νέους στην ελλάδα και να βοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή χρειάζονται νέοι πόροι. Ε, και θα ήθελα να παρακαλέσω να κοιτάξουμε τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα με μια συνοχή ως προς τις άλλες πολιτικές, δηλαδή την κοινωνική συνοχή και την ε, οικονομία, ιδιαίτερα την πράσινη οικονομία. Σας ευχαριστώ. Ματίας, ε, για ένα λεπτό. Κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επαναπρογραμματίσουν τα εθνικά ταμεία για να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Πέρσι, το τέλος του παρελθόντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει τη διάθεση διεθνωτικών πόρων στις χώρες εκείνες που δεν συμμορφωνόταν με τους στόχους που είχαν τεθεί όσον αφορά την μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυής για να καταλάβει ότι, ότι αυτό αποτελούσε απειλή και τιμωρία. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Επίτροπο. Η απόφαση αναστολής διαθέσεως των διευθυντικών πόρων όταν δεν πληρούνται οι στόχοι για το δημοσιονομικό έλλειμμα, εξακολουθεί να ισχύει αυτή η απειλή. Εν τη αυτή περιπτώσει η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα διαθεωτικά ταμεία, θα έχουν δικαίωμα, αν αρθεί αυτή η απειλή. Μπορεί να μας δώσει μια άμεση απάντηση σε αυτό σας παρακαλώ, διότι έχουμε κουραστεί από αυτές τις ε, απειλές και, τις, ε, και τρομοκρατίας στην ε, Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Τεϊσέρα για 1,5 λεπτό. Κύριε Τεϊσέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, σύμφωνα με τη Eurostat, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση έχει περίπου 23 εκατομμύρια ανέργους. Αυτό είναι 3% πάνω από το 2008. Κυρίως οι νέοι δεν βρίσκουν θέσεις στην αγορά εργασίας η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 20%. Στην Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι 19% και 17% στην Ιαπωνία. Θα πρέπει να τονώσουμε λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε πλούτο και να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Τα 82 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα μόνο 3 δισεκατομμύρια προορίζονται για την Πορτογαλία. 14% του ποσού από το 2011 μέχρι το 2014. Δεν έχουν διατεθεί σωστά στην Πορτογαλία. Χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά για να δώσουμε κάποιο δυναμισμό στην οικονομία μας, για να υποστηρίξουμε μικρές επιχειρήσεις, να υποστηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και να υποστηρίξουμε το τουρισμό μας και να δημιουργήσουμε θέσεις για τους νέους. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για να προωθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε θέση για του νέου για να ανταποκριθούμε στι ανάγκε τη αγορά εργασία. Θα ήθελα να ρωτήσω τι συγκεκριμένα μέτρα ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται αυτές τις συμβουλές διότι η Πορτογαλία θέλει να φύγει από τη λιτότητα προς την οικονομική ανάπτυξη για να δημιουργήσουμε πλούτο και θέσεις απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τι ερχολέν για ένα λεπτό. Κύριε Επιτροπέ, η πρωτοβουλία αυτή καλές προθέσεις έχει. Πρέπει να είναι αυτές οι προτεραιότητές μας ε, μεταξύ άλλων απασχολησιμότητα των νέων, αλλά και η επένδυση στο μέλλον. Θέλουμε να διατηρήσουμε μια δυναμική και μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά σε ό,τι αφορά ε, την ε, συνοχή της πολιτικής, τη συνεκτικότητα της πολιτικής, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Αν προχωρήσει σε μια στήρα λιτότητα, λιτότητα για τη λιτότητα ως αυτός σκοπός, τότε δεν θα υπάρξει ανάπτυξη ούτε για τις μικροψηφίες επιχειρήσεις, ούτε θέσεις εργασίας για τους νέους και θα έχουν χαθεί άδικα όλοι μας οι κόποι. Πώς εξηγείτε επίσης κύριε Επίτροπε την πρότασή σας να μειώσετε κατά περίπου 50% κάποια ταμεία για τις άκρος ε, απόκεντρες περιφέρειες όπου η ανεργία των νόμων πολλές φορές περνά και το 60%. Είχατε όμως δεσμευτεί να διατηρήσετε αυτές τις περιφέρειες που όμως τελικά τιμωρούνται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Πού είναι η δικαιοσύνη λοιπόν, πού είναι η συνεκτικότητα. Η απόφαση αυτή λοιπόν δεν είναι δυνατόν να τύχει τη υποστήριξή μας. Είναι απαράδεκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Καντέκ για Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω πόσο ωραία νιώθουμε στο Στρασβούργο. Το λέω έτσι για να μην το ξεχνάμε, κάθε φορά θα το λέω. Η πρόταση Μπαρόζο έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Αναθρωτικών Ταμείων έχει στη διάθεσή της ένα δημόσιο μέσο επενδύσεων πολύ σημαντικό δύσκολη καιρή για τις οικονομίες των κράτων μελών, αλλά πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Με βάση τον πρόεδρο της Κομισιόν, 82 δις ε, ευρώ τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί το 2007 στο 2013 θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν υπέρ των νέων κατά της ανεργίας τους. Ε, Τρέφομαι λοιπόν ε, και ρωτώ πού είναι αυτά τα κονδύλια. Ήταν κονδύλια τα οποία δεν είχαν προγραμματιστεί μέχρι τώρα είχαν διατεθεί για τα κράτη-μέλη και ήταν για επιχειρησιακά προγράμματα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επαναπρογραμματιστούν τα κονδύλια αυτά, διότι αυτό μπορεί να ε, μην έχει τελικά ευεργετικές επιπτώσεις επιτόπου. Να πω δε ότι ήδη τα διαθωτικά ταμεία ε, βοηθούν και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και του νέου. Αλλά σίγουρα αυτά πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και για το μέλλον, το μελλοντικό προγραμματισμό. Ο πρόεδρος Σαρκοζή αποφάσισε να εφαρμόσει το φόρο ε, στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ε, το λέω στον συνάδελφο που κάτι είπε πριν, μήπως και δεν το έχει λάβει υπόψη του, τον κύριο Μπεζέ. Σας ευχαριστώ. Μπαζέσκου για 1,5 λεπτό, κυρία Μπαζέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την παρούσα κρίση αν δεν καταφέρει να υποστηρίξει τους νέους της, ούτω ώστε να μπορέσουν να βρουν θέσεις απασχόλησης, τις οποίες δημιουργούν οι επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε να δώσουμε δουλειά στους νέους για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν το συνταξιδοτικό σύστημα που, μιας Ευρώπης που γυράσκει. Τα στοιχεία που μας έδωσε η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης των νέων στη Ρουμανία, πάνω από 100.000 νέοι κάτω από τους 30-30 ετών βρίσκονται στην ανεργία. Οι πιο μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζονται στην πρώτη θέση εργασίας. Το κράτος της Ρουμανίας δαπανά πάνω από 1,17 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο Γι' αυτό κάθε μορφή χρηματοδοτήσεως και υποστηρίξεως για τους νέους επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει κατά πόσο έχει την πρόθεση να μειώσει τα ποσά που διατίθεται στις χώρες εκείνες που έχουν επίπεδο απορροφήσεως χαμηλό Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτέ οι χώρε ακριβώ είναι αυτέ που πρέπει να υποστηριχθούν ούτως ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα χρήσεω των ευρωπαϊκών πόρων. Η μείωση του ποσοστού τη χρηματοδότηση ήταν μια δυνατότητα για αυτό το σκοπό. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δώσει ένα σχέδιο δράσεω για τη χρήση των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε προγράμματα μαθητείας και κατάρτιση. Υπογραμμίζω ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η μεθοδολογία, ούτω ώστε να προσφέρονται τα απαραίτητα εχέγγια για την χρηματοδότηση των νέων επιχειρηματιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη πρόκληση για μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για τους νέους σε όλη την Ευρώπη. Επίσης και άλλο θέμα είναι να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη εν γέννη εάν θέλουμε να το πετύχουμε, μάλλον το πετύχουμε αυτό θα είναι καλό. Θα πρέπει τώρα το να μεταφερθούν πόροι από τα διευθυντικά ταμεία και να διατεθούν και να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται μια πρακτική διευθέτηση. Και πρόσεξε αυτό που έθεσε η κυρία Ένστ για την Ιρλανδία, όπου η χώρα ήδη χρησιμοποίησε τα διευθυντικά ταμεία, τα διευθυντικού πόρου. Πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. παρόλα αυτά, στο ότι αυτό μπορεί να γίνει νομίζω ότι 82 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα, 3 δισεκατομμύρια ανακάτως μέλος και μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Αλλά α υποθέσουμε ότι μπορεί να συμβεί. Ζητώ κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται κάποια ευελιξία. Διότι αν δεν υπάρχει ευελιξία, βλέπω ότι οι κατοικοί φορεί να καταπίνουν τα χρήματα και να μην είναι ω αποτελεσματική χρήση του όσο θα έπρεπε. Ο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μπορέσει να συμμετάσχει και από πλευρά παιδεία, κατάρτιση και δημιουργία ε, ευκαιριών. Και η κατάρτιση θα πρέπει να βασίζεται πρακτική προσεγγίσεω. Να μην είναι κάτι τυπικό, γενικό, αυτά που μας δίνουν κρατικοί φορείς συνήθω και το λέω αυτό ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τα, τη χρήση των πόρων στην Ιρλανδία και θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των διαφόρων φορέων τοπικών και των νέων ότι αυτό μπορείτε να συμβεί, να το χρησιμοποιήσουν και να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Αν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, μπορεί πραγματικά να κάνουμε κάτι, να κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, κύριο Λαβία έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ε, κυρία Προέδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, τα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, συζητούν τις κατευθύνσεις για τον προπολογισμό του 2013 και οι συζητήσεις έδειξαν ότι υπάρχει συντονισμός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν όσον αφορά την πολιτική δράση της Ένωσης. Συγκλίνουν επί της ανάγκης να προωθηθεί η ανάπτυξη και μέσω της καταπολεμήσεως της ανεργίας, κυρίως ε, την ανεργία των νέων θέλουν να καταπολεμήσουν. Δέχομαι γι' αυτό πολύ καλά τη διακήρυξη για τη χρήση των 82 δισεκατομμυρίων ευρώ του προγραμματισμού 2007-2013 υπέρ των μικρομεσών επιχειρήσεων που είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας. Όπως απεδείχθηκε από στατιστικές που έδωσε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλουμε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει το 85% των θέσεων εργασία που δημιουργήθηκαν από το 2002 μέχρι το 2010. Ε, πιστεύω ότι είναι προφανή η ανάγκη να γίνει μια κοινή προσπάθεια με μια οπτική συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ ευρωπαϊκών προπολογισμών και εθνικών προπολογισμών για να εστιαστούν οι πόροι και να επαναπροσελιστούν οι πόροι των κρατών μελών υπέρ των προτεραιοτήτων που εξεφράστησαν και πιο συγκεκριμένα προ τα μέτρα εκείνα και τα προγράμματα εκείνα που είναι σε θέση να, έχουν, να επηρεάσουν και να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα και να αντιστραφεί η ρότα που ακολουθούν οι νέε σε αυτή τη φάση. Ζητώ από τον Επίτροπο να ξεκαθαρίσει τι δράσει, τα προγράμματα και τα κονδύλια του προπολογισμού ε, και εκείνα που θα διατεθούν τα ποσά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την καινοτομία. Πώ μπορούν να ενισχυθούν τα ποσά για να μειωθεί η ανεργία των νέων. Μπορεί να το ξεκαθαρίσει, να δώσει περισσότερε λεπτομέρειε ο Επίτροπο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο Νικολέσκου, για ένα μισή λεπτό. Κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν είναι γενναιόδορη και Φαντάζομαι καλοπροαίρετη. Αλλά μας λέει ότι πρόκειται για πόρους οι οποίοι πηγαίνουν ε, σε σχέδια μεγάλης εμβέλειας, σχέδια υποδομών. Και κάποιοι από αυτούς τους πόρους, με άλλο μέρος τους, πηγαίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους νέους. Καλή αυτή η κατανομή. Θα μπορούσε να ωφελήσει τα κράτη-μέλη που θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στους δύο αυτούς τομείς. Αλλά η επιλογή θα πρέπει να γίνει ατομικά από κάθε κράτος μέλος, ξεχωριστά. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον επαναπρογραμματισμό εσωτερικά των προτεραιοτήτων. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ευρωπαϊκών Ταμείων είναι η έλλειψη πόρων για την εθνική συγχρηματοδότηση και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Higgins, ο κύριος Higgins έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα συγχαρώ την κυρία Χίπνερ για την επίκαιρη προφορική ερώτηση. Η οικονομική κρίση έχει ρημάξει την απασχόληση των νέων. Τα στατιστικά στοιχεία είναι τρομακτικά. Μιλάμε για λιγότερο από 10% ανεργία των νέων μόνο σε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία. Αλλού είναι δραματική η κατάσταση. Βαλτικέ χώρες, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ελλάδα. Μιλάμε για ανεργία νέων 30% και πάνω. Στην Ισπανία δεν πάνω από 40%. Μιλάμε για διαφυγή εγκεφάλων που δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε. Χρειαζόμαστε νέους εργαζόμενους για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση που αντιμετωπίζουμε από τι οικονομίε χαμηλού κόστου. Άρα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε στους νέου μα. Είναι νέοι, έξυπνοι, πολλοί από αυτού με προσόντα, αλλά είναι να μείνουν στη χώρα μα και μιλάω, βλέπω και τη δική μου τη χώρα που ευτυχώ βγαίνουμε από την οικονομική κρίση, πολλοί από αυτού με τριτοβάθμια πτυχία, με διδακτορικά, φύγανε στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε πολλέ περιπτώσει δεν θα επιστρέψουν. Λόγια ακούσαμε πάρα πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, σημαντικές, στη χώρα μου είναι 60% της απασχόλησης, αλλά συμφωνώ με τον συνάδελφό μου τον Σον Κέλλη. Εάν είναι να έχουμε ευέλικτα συστήματα, δεν θα πρέπει να έχουμε γραφειοκρατία. Πάρα πολλά εξαιρετικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άκαμπτα και γραφειοκρατικά και δεν λειτουργούν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ερώτηση που συζητούμε απόψε είναι ύψιστη σημασία σημασίας γιατί αναφέρεται στου νέου, το σπουδαιότερο κεφάλαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλήττεται σήμερα από ανεργία και ανασφάλεια όχι μόνο στι χώρε με τα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα όπω είναι η χώρα μου η Ελλάδα αλλά και σε άλλε χώρε του Βορρά και του Νότου. Οι νέοι αναγκάζονται να εκπατριστούν και όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και εκτό Ευρώπη. Ο προσανατολισμός προ την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη μέθοδος διότι οι επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν τα ταλέντα των νέων με τις καινοτόμες ιδέες με την υψηλή εκπαίδευση που έχουν οι ευρωπαίοι νέοι αλλά μπορούν να αποτελούν και ένα αντικείμενο δικής τους δημιουργίας. Ε, τα διαφορετικά ταμεία οφείλουν να συμβάλλουν σε αυτή την περίπτωση είναι το βασικότερο εργαλείο που έχουμε σε μια ευρώπη που στερείται μηχανισμών αλληλεγγύης και άμεσης αντίδρασης στην κρίση και στην επίλυση των προβλημάτων. θέλω κάποιες ερωτήσεις να θέσω κύριε επίτροπε. τα 82 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επενδυθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα συνοδεύονται μέσα από τα σχέδια δράσης και από συμπληρωματικές πολιτικές. πολλές φορές τα εμπόδια δεν είναι η έλλειψη πόρων αλλά είναι διοικητικά είναι νομοθετικά ε, χρειάζεται και επένδυση σε τομείς συμπληρωματικούς όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας η καινοτομία. θα ήθελα επίσης να ρωτήσω θα συνοδευτούν και από ευελιξία αυτή η νέα κατεύθυνση των πόρων. Ε, υπάρχουν περιοχές που έχουν έντονα διαρθρωτικά προβλήματα και θέλουν άμεσα λύσεις σωστά σχεδιασμένες και επικεντρωμένες στα προβλήματά τους. άλλες που πλήττονται από έκτακτες καταστροφές. στη χώρα μου στην ελλάδα η ηλία μια ειδική περιοχή θα μπορούσε να ωφεληθεί από ένα τέτοιο πρόγραμμα με ευελιξία και αμεσότητα. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν δέκα αιτήματα για αγόρευση σύμφωνα τη διαδικασία Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο σε όλους. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο που σας διατίθεται. Ο κ. Νικολάζικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η πρόταση του κυρίου Μπαρόσο για να πάνε τα διάθετα κονδύλια στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις όλα αυτά οδηγούν σε κάποιες αμφιβολίες και ανασφάλειες στα κράτη-μέλη όσον αφορά την αναγκαιότητα βεβαίως του βήματος αυτού. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος ε, σημαίνει το εξή ε, για την περίοδο 2007-2013 υπάρχει απορρόφηση μέχρι στιγμής μόνο του ενός τρίτου των κονδυλίων αλλά ακριβώς υπάρχει μια μεγαλύτερη επιτάχυνση στο τέλος της ε, προγραμματικής περίοδου και υπάρχει ο κίνδυνος να μην επαρκέσουν τα κονδύλια για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και να χρησιμοποιηθούν ε, τελικά άσκοπα. Ευχαριστώ, Λουκατσεύσκα. Κύριε Λουκατσεύσκα, έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου, δεν την ακούν οι διερμηνείς, δυστυχώς. Słychać? Σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, παίρνω για δεύτερη φορά το λόγο, διότι πολύ με προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα της κατάρτισης. Πάρα πολλά χρήματα δαπανώνται για μη επαρκή κατάρτιση στατιστικά. Είναι καλά τα στοιχεία, χρησιμοποιούνται οι πόροι, οι εταιρείε που δίνουν την κατάρτιση είναι ικανοποιημένε, διότι αυτοί που εργάζονται για αυτού μπορούν να έχουν τη θέση του ε, διότι πρέπει να καταρτιστούν οι άνεργοι και ε, ενθαρρύνονται και από κάποια οικονομικά κίνητρα για να συμμετάσχουν στην κατάρτιση αλλά δεν μπαίνουν στην αγορά εργασία αυτά που έχουν υποστεί την κατάρτιση. Αυτή η κατάρτιση είναι αυτό σκοπός. Δεν δίνει τι αναγκαίε δεξιότητε στο εργατικό δυναμικό για να απορροφηθεί. Το ερώτημά μου, Επίτροπε, μπορείτε να μα πείτε κατά πόσο έχουν γίνει κάποιε μελέτε, πόσο κοστίζει να επιστρέψει ένας άνεργος στην αγορά εργασίας και ποιο ποσοστό τον πόρων που διατίθεται από τις ευρωπαϊκές πηγές ε, πηγαίνουν για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η κυρία Μπερέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτροπέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση έρχεται ως αντιστάθμιση, ως αντίβαρο στον λεγόμενο χρυσό κανόνα που εγκρίθηκε. Η νέα συνθήκη ε, δεν έχει καμία διάταξη υπέρ της ανάπτυξης και της απασχολής, άρα καλό είναι και αυτό. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε μια συνθήκη και από την άλλη πλευρά τη δήλωση αυτή που πρέπει να φέρεται σε πέρας σήμερα. Καλές ιδέες ε, ε, θα χρειαστείτε για να προωθήσετε την απασχόληση των νέων. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να, να δείτε τις εργασίες του Κοινοβουλίου μας, διότι εμείς εκπονήσαμε μία έκθεση για την απασχόληση των νέων και πιστεύω σε αυτήν την έκθεση θα βρείτε καλές προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρησιμοποίηση των πόρων των ενθρωτικών ταμείων, βλέπουμε πάρα πολλές μεγάλες, πολύ μεγάλες αντιφάσεις ε, στο σώμα των επιτρόπων όταν πρέπει να σταθμίσουν ε, τον ε, χρυσό κανόνα, λένε κινητοποίηση των ανθρωπτικών ταμείων. Αλλά από την άλλη πλευρά ε, τιμωρούνται τα κράτη-μέλη τελικά. Και κάποια στιγμή πρέπει να επιλέξετε. Τι πολιτική θα ακολουθήσει ώστε να είστε Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί μπορώντας να στηριχθεί και στα δυο της πόδια. Και σε ό,τι αφορά και τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, αν δούμε την πρόταση Μπαρόσο, έχουμε κάποια ερωτηματικά. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μπορεί να έχει πόρου που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν ανάλογα με τη συγκυρία για να υλοποιηθούν αντικυκλικά μέτρα. Οι προτάσεις που κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση για το μελλοντικό σχήμα των εθνικών ταμείων είναι προσαρμοσμένα στην κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κατάσταση κρίσης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε το Μάρτιο να δώσει κάποιους προσανατολισμούς ε, όσον αφορά την απασχόληση στα κράτη-μέλη, ε, τονίζοντας την ανάπτυξη και την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας. Είναι σημαντικό να γίνει σωστός αναπρογραμματισμός των θετικών ταμείων προς καλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη απασχόληση πρέπει αυτά να γίνουν εντός ε, του πλαισίου που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος μέλος. Τα κάτι μελη πρέπει να διαθέσουν πόρους για να τονώσουν την απασχόληση, κυρίως αυτή των νέων, και για να τονώσουν τη λειτουργία της οικονομίας και πάνω απ' όλα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να υποστηριχθούν πάνω απ' όλα τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να ρυθμίσουν τα οικονομικά τους. Διότι αυτές τις χώρες η οικονομική κρίση έχει επιφέρει και κοινωνική κρίση πάρα πολύ ε, εμφανή. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι δεν παίρνουν κανένα επίδομα ανεργίας και ούτε άλλη μορφή κοινωνικής ενίσχυσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε στο δίκτυο το επίπεδο απασχόλησης και όχι αυτό της ανεργίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Φερέιρα. Κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι ανακοινώσει που έγιναν όσον αφορά τον αναπρογραμματισμό των θετικών ταμείων χρήζουν διευκρινήσεων. Είναι μια ρητορική αυτή που ακούγεται, προσπαθεί να καλύψει τα καταστροφικά αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιανουαρίου. Το να μιλάμε στην ίδια συνεδρίαση για ανάπτυξη και απασχόληση, στην ίδια συνεδρίαση που θέσπισε μέτρα λιτότητας ε, και που ζήτησε περισσότερη φιλελευθερωποίηση και που επετέθη κατά των νόμων μας περί εργασίας ε, και οδήγησε απολύσεις δεν είναι ε, ρητορική αλλά το αποκορύφωμα της υποκρισίας. Είπε ο πρόεδρο τη ότι μπορούσαν να δετεθούν σε όλα τα κάτι μελη 82 δισεκατομμύρια του ποσού στα κάτι μελη 40, 42 χρειάζεται ο λαός της Πορτογαλίας να πληρώσει τους τόκους ε, που οφείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Δούνου του. Αντί να γίνει επαναπρογραμματισμό, αυτό που χρειάζεται είναι μια ουσιαστική αύξηση των διχοδοτικών ταμείων, των, των πόρων του, ώστε να συνεργαστούμε μέσα σε αλληλεγγύη και να μην πρέπει να ακούμε προσβλητική προπαγάνδα. Χρειάζεται να τεθεί τέρμα σε αυτή την, ε, ε αυτόν τον εκβιασμό και την πολιτική που ασκείται που αυξάνει σε, α, πρωτοφανή επίπεδα την ανεργία και που πνίγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πολιτική που ακολουθείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάσκα. Κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι νέοι χρειάζονται δουλειά και οι πολιτικοί ακολουθούν. Ε, χαιρετίζω λοιπόν την αντίδραση της ε, Κομισιόν σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχει ανέβει πάρα πολύ η ανεργία των νέων. Η πρόταση να χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η εργασία των νέων με αδιάθετα κονδύλια είναι πάρα πολύ θετική. Σε δύο δε χώρες πλησιάζει το 50% η ενεργεία των νέων και σε άλλες είναι πάνω από το 30%. Οι νέοι λοιπόν μετά από ένα διάστημα ανεργίας σταματάνε να αναζητούν εργασία και το μόνο εισόδημα είναι τα κοινωνικά επιδόματα. Γι' αυτό χαιρετίζω την ε, πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν ε, να συνδέσει την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την απασχόληση των νέων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ματούλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση του Πρόεδρου Μπαρόζο έχει ως στόχο την άρση του οικονομικού αδιεξόδου με την εφαρμογή μέτρων τα οποία στόχο έχουν την δρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μείωση της ανεργίας των νέων. Όμως, η αλλαγή του επιμερισμού των ποσών που δεν δαπανήθηκαν θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τη συνθήκη και την ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι αρμοδιότητες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ απλό το θέμα τελικά. Μπορεί ένα κράτο μέλος να χάσει ε, τους πόρου πόρους από τα διαδροτικά ταμεία στα, τα οποία δικαιούτο με αυτήν τη νέα κατανομή. Στόχος είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις στις, και οι στέρησεις στις περιφέρειες. Θα μπορούσαν να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από τα αποτελέσματα, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει περισσότερες ε, διευκρινήσεις ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή αυτής της πρότασης ε, του κ. Μπαρόζο, αλλά και σε ό,τι αφορά το σεβασμό του βασικού στόχου της πολιτικής συνοχής. Ο επαναπρογραμματισμό λοιπόν των 82 δι θα πρέπει να λάβει υπόψη μια καλύτερη ευελιξία, μια πιο εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και βελτίωση ε, τη διοικητική ικανότητα των δικαιούχων. Ευχαριστώ. Άλβες. Κύριος Άλβες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρόταση του Πρόεδρου Μπαρόζο για τον επαναπρογραμματισμό των διαθέσιμων κονδυλίων που θα στηρίξουν τελικά την ε, απασχόληση ιδίω των νέων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Έρχεται στην κατάλληλη χρονική στιγμή, ιδίω για τις χώρες ε, που υφίστανται μέτρα λιτότητας, όπως η Πορτογαλία με τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες χρηματοδότησης οικονομίας και δι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν ε, μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από τις τράπεζες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να διατεθούν πόροι στις περιφέρειες και ιδίως στις αζόρε με πάρα πολύ, μεγάλο, πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας. Μιλάμε για ύφεση, έχουμε πολύ μεγάλη ύφεση σε διεθνέ επίπεδο. Μας προτείνεται τώρα μία διέξοδο με αυτά τα διαρθρωτικά κονδύλια. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους. Νέους πολύ καλά εκπαιδευμένους, μορφωμένους, με προσόντα που δυσκολεύονται να βρουν μια θέση εργασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ξέρω είναι πώ θα εξασφαλιστεί στην πράξη η πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και πώ θα συμμετάσχουν στον επαναπρογραμματισμό οι περιφέρειε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ρέγνερ. Κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Επίτροπε. Δεδομένου του σκότους της λιτότητας, τα μέτρα αυτά χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων είναι πάρα πολύ αναγκαία. Είμαι από την Αυστρία και ξέρετε πόσο ο επικεφαλής της ε, κυβέρνησής μας παρουσίασε την πρόταση για τους νέους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, δόξα τω Θεώ, η ανεργία των νέων χαμηλή στην χώρα μας. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει διπλή κατεύθυνση στην εκπαίδευση από πάρα πολύ νωρί και βέβαια όλοι γνωρίζουν πώς έχουν μια θέση η εκπαίδευση ή η κατάρτιση και θα πρέπει να υπάρξει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι πάρα πολύ σωστά όπως λέτε μια ανάλογη εγγύηση σε ευρωπαϊκή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω μπορούμε να δημιουργήσουμε τα 2 εκατομμύρια, 2 θέσεις, 2 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τους νέους με το απλοποιημένε διαδικασίες και το ποστό χρηματοδότησης 10% αλλά θα ήθελα να προσέξετε να μην πάνε από τη μία τσέπη στην άλλη μόνο τα λεφτά κύριε Επιτροπέ. Τελευταία παρέμβαση. Πρέντελ Γκάστ. Κυρία Πρέντελ Γκάστ. Ευχαριστώ πολύ. Η αδίποτε δήλωση στο άτυπο Συμβούλιο τη περασμένη εβδομάδα, σε μια δήλωση του κ. Μπαρόσο, εισήγαγε την έννοια των ομάδων δράση που θα κινούνται στο τοπικό επίπεδο για να καταπολεμήσουν την ενεργεία των νέων. Οι ομάδε δράση θα δημιουργηθούν στα 8 κράτη μέλη σε δυσχερή θέση. Συμπληρώνεται η Ιρλανδία σε πιλωτική βάση και διερευνηθούν τρόποι χρήσεω των πόρων που θα μπορούσαν να προγραμματιστούν από τα περιφερειακά ταμεία και τα εθνικά ταμεία του κράτου μέλου αυτού για προγράμματα για την ανακούφιση τη ενεργεία των νέων. Δεν μπορούμε να κάνουμε περικοπέ από τα προγράμματα εθνικών ταμείων για να εισαγάγουμε νέα προγράμματα. Χρειαζόμαστε συμπληρωματική χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Χρειαζόμαστε σίγουρα συμπληρωματικά μέτρα και η οικονομική διακυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη για να βοηθήσουμε να μειωθεί το βάρο τη ανεργία των νέων και να εξασφαλίσουμε ότι τη νέα γενιά δεν θα έχει υπερβολικό βάρος στους ώμους της από αυτή την κρίση και ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε παιδεία, κατάρτιση και απασχόληση. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση έδειξε πως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει πάρα πολύ καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων, κάτι το οποίο βεβαίω είναι αναμενόμενο και ευχάριστο για τον αρμόδιο επίτροπο. Αλλά βεβαίω η συζήτηση δείχνει, κάτι που είναι σαφές, πως τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένα μέσο πολύ αποτελεσματικό που καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη για να επιτύχουμε ευρωπαϊκούς στόχους. Θα ήθελα να δείτε την πρόταση του Πρόεδρου Μπαρόζο, κυρίες και κύριοι, ως ένα ξύπνημα όσον αφορά την έφλεκτη και εμπριστική κατάσταση στο πλαίσιο της ανεργίας των νέων. Βεβαίως είναι προφανές ότι γνωρίζει τους κανόνες λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλά ήθελε να δηλώσει πως αυτή την στιγμή ένα από 82 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένα έργα και είναι θεμητό να αναρωτηθεί κανείς εάν υπάρχουν οι δυνατότητες μήπως μπορεί να ανακατανεμηθεί όχι προφανώς σε ε, έργα άλλα, αλλά μέσω μετακίνησης εντός των περιφερειών με βέλτιστη στοχοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης των νέων. Μην ξεχνάμε πως τα επιχειρησιακά προγράμματα το 2005-2006 είχαν συζητηθεί, συμφωνηθεί και εγκριθεί σε τελείως διαφορετικό οικονομικό κλίμα. Γι' αυτό είναι σωστό να θέσουμε το ερώτημα εάν μπορούμε τώρα στοχευμένα να ξαναδούμε την κατάσταση. Αυτό έκανε η Κομισιόν και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στις 8 χώρες με την υψηλότερη ανεργία των νέων αναλαμβάνουμε δράση να μιλήσουμε με τους αρμόδιους των κρατών μελών για το να δούμε τι μπορεί να γίνει και από πλευράς Κομισιόν αρχές Μαρτίου θα ε, σας δώσουμε μια πρώτη προφορική αναφορά αυτών των συζητήσεων αλλά σας διαβεβαιώ ήδη πως ο συνάδελφός μας, ο κύριος Άντορ, κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε την προεργασία για το θέμα αυτό, για τις ευκαιρίες των νέων. Με στόχο να γίνουν προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει στην ανεργία των νέων. Και ακριβώς αυτές οι προτάσεις τώρα θα ενσωματωθούν στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για να εφαρμοστούν, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις κατά περιφέρεια και πιθανώς κάτω από το επίπεδο της περιφέρειας κιόλας για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά νομίζω δίκαιο είναι να πούμε πως ούτε και εδώ πέρα από τη μια μέρα στην άλλη θα έχουμε μια δραματική βελτίωση της κατάστασης. Αλλά ποιο είναι το θέμα και εδώ πέρα συμφωνώ οπωσδήποτε με την έκκληση του Πρόεδρου της Κομισιόν πρέπει να δράσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να λάβουμε την πρωτοβουλία και ελπίζω όλοι να έχουμε τον ίδιο στόχο. Και είμαι πεπισμένο πως ήδη σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα πρώτα τα αποτελέσματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Τώρα ερχόμαστε στις παρεμβάσεις της